Siamo in attesa dell'onorevole Nibler e quindi dobbiamo attendere qualche secondo. Αναμένουμε τώρα την κυρία Νίμπλερ, η οποία είναι καθοδόν. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε δυστυχώ τη μερίσια διάταξη, οπότε θα πρέπει να σταματήσουμε για πέντε λεπτά. Ε, ε και λιγότερο. Θα περιμένουμε την κυρία Νίμπλε. Βρίσκεται καθοδόν, σα είπα. Επανερχόμαστε στην έκθεση Νίμπλερ για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανία. Αν είναι έτοιμη η κυρία Νίμπλερ θα της δώσω το λόγο. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητής Συνα... Αγαπητή κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, πολλές γερμανικές εφημερίδες αναφέρουν ότι το EADS θα αναγκαστεί να απολύσει πολύ κόσμο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και διαστημικής βιομηχανίας. Πολύ, πολλά εργοστάσια θα κλείσουν και αυτό προσωρινά τουλάχιστον και κινδυνεύουν πολλές ε, ε θέσεις εργασίας. Η διαστημική βιομηχανία ε, καλύπτει το 1 τρίτο των εργαζομένων του ΕΑΝΤΕΑΣ στην Βαβαλία, στη Βαβαρία. Οι βιομηχανικές ε, δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με και οι άλλες ε, εργασίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι μεγάλη σημασία και για τον πολιτικό τομέα. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να κερδίσουν πολλά από τα προϊόντα που είναι αποτελέσματα της διαστημικής έρευνας και αυτό αυξάνει την ευμάρεια των πολιτών μας και μπορούμε όλοι να έχουμε άμεσα ή έμεσα ωφέλη από τη δημοσιακή ε, βιομηχανία. Παραδείγματος χάρη τηλεόραση, το ίντερνετ μεγάλης ταχύτητος, το, τα συστήματα πλοήγησης κτλ. Και ακόμα και η γεωργία ευνοείται από την δυνατότητα τηλεεπισκόψη. Είναι όμως απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τα βασικά προβλήματα του διαστημικού κλάδου που είναι η χρηματοδότηση. Είναι μια βιομηχανία που έχει μεγάλη ένταση χρηματοδότηση με μακρούς κύκλους ανάπτυξης. Είναι η ασφάλεια των επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα. Είναι πολλά χρήματα τα οποία επενδύονται στην καινοτομία όταν δεν είναι σίγουρο αν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα αγοράσει το προϊόν τους. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αρχική ε, χρηματοδότηση συρμαγιάς για τις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες θέσεις απασχόλησης και να προχωρήσουν σε αυτή την έρευνα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια συνεργασία για την ευρωπαϊκή ε, πολιτική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΖΑ και των κρατών μελών, που να καλύψει και το χρονικό διάστημα μέχρι το 2020. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να είναι και η βάση τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα έχει το λύσει στην ανάγκη να υπάρξει μια φιλόδοξη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα και πρέπει να το τονίσουμε και πάλι. Ο Γαλιλαίο ε, είναι απαραίτητο να περατωθεί το ταχύτερο δυνατόν ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα ωφέλη που προσποριζόμαστε από αυτό, όπως παραδείγματος οι επικοινωνίε μέσω δορυφόρου. Ε, είναι απαραίτητο επίσης να αποκτήσουμε και μια ανεξαρτησία από άλλους ε, από άλλες οντότητες οι οποίες ε, έχουν διαστημική δύναμη. Έτσι μονάχα μπορούμε να κρατήσουμε τις εχώριες βιομηχανίες μας και την ανταγωνιστικότητά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κέλλη. Φαντάζομαι ότι το διάστημα είναι ένα θέμα το οποίο μαγεύει πολύ κόσμο, αλλά φαίνεται ότι αυτή η μαγεία δεν ε, βρίσκει συγκεκριμένη έτσι, ε, ε, πνοή στην βιομηχανία η συνάδελφος Νίμπλερ μόλις ε, αναφέρθηκε στο μεγάλο δυναμικό που ε, υπάρχει στην ε, βιομηχανία αυτή. Βεβαίω εδώ και χρόνια έχουμε προβλήματα με τον Κοπέρνικο, με τον Γαλιλαίο. Πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουμε περισσότερο και ενδεχομένως θα πρέπει να δούμε τι κάνουν και η Κίνα, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε που φαίνεται ότι βρίσκονται όλοι μπροστά από μας. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την εσωτερική αγορά όσον αφορά την διαστημική βιομηχανία, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. Εταιρείε, ε, οι οποίες ε, έρχονται από όλο το φάσμα ε, της διαστημικής βιομηχανία έχουν αυτή αυτά τα συστήματα, τα τα τριμετρικά, τα οποία ε, μπορούν ε, να δώσουν λύσεις σε προβλήματα ε, πολύ πιο συγκεκριμένα, όπως ας πούμε να απομονώσουν δάση, αλλά ακόμα και με μονομένα δέντρα, το μέγεθός τους που βρίσκονται, πώς μπορεί κανείς να τα βρει κτλ. Και, και νομίζουμε ότι αυτό δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες ε, στην ε, βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σόλτ. Η τεχνολογία αυτή έχει αναπτυχθεί σε τμήματα της ε, δικής μου εκλογικής περιφέρειας που επιτρέπει την παρακολούθηση του ηλίου, του γαλαξία και ακόμα και επαλήθευση της θεωρίας του Αϊνστάιν. Τα συστήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και φυσικά χρειάζονται την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλουμε να κερδίσουμε το νέο αγώνα στο διάστημα για τεχνολογία και θέσεις απασχόλησης. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Νίμπλερ και πράγματι και εγώ ανησυχώ μετά από την ανακοίνωση της ΕΑΝΤΕΕΣ σε σχέση με τη διαστημική και αμυντική δραστηριότητά τους αλλά ε, χαίρομαι που το Ηνωμένο Βασίλειο και η εγκαταστάσει εκεί του ΕΑΝΤΕΣ θα παραμείνουν τμήμα του πυρήνα των δραστηριοτήτων και η εταιρεία θα κάνει τις ε, απώλειες θέσεων απασχόλησης με τη φυσική αποχώρηση των εργαζομένων και όχι με απολύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν μια δυσμενή κατάσταση στον εργασιακό κόσμο. κύριος Κουρέα. Κυρία Πρόεδρε, θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και να πω την απαραίτητη μια πολιτική στον διαστομικό τομέα η οποία να έχει σταθερότητα και ικανότητα ανταγωνισμού με τους άλλους μεγάλους παγκόσμιους εταίρους με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΣΑ και των κρατών μελών. Ο Γαλιλαίος, ο Κοπέρνικος, ο Έγνος είναι οι προτεραιότητέ μα πρέπει να καλύψουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι τα βέλτιστα παραδείγματα μια διαστημική πολιτική συνεκτικής και ανταγωνιστικής με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλη έμφαση επίσης στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το ρόλο της διαστημικής βιομηχανίας ως φορέα καινοτομία και ανάπτυξη. Είναι ένα σημαντικό τομέα για την ασφάλεια των πολιτών για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κρίσης για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας, για την καθημερινή ζωή με τι μεταφορές και τις επικοινωνίες, ένα τομέα ο οποίο απαιτεί πιο έντονες ε, και μεγαλύτερη όθηση. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Νίμπλερ, την εισηγήτρια, για αυτή την ε, τόσο ε, ενδιαφέρουσα και σημαντική έκθεσή της, για αυτή την τόσο σημαντική ε, βιομηχανία. Είναι μια βιομηχανία η οποία δημιουργεί τεχνολογική καινοτομία και αυξάνει την τεχνογνωσία της Ευρώπης άλλωστε έχουν δεσμευτεί πολλά εκατομμύρια ευρώ στο επόμενο δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο για την έρευνα και για τον ε, Γαλιλαίο. Ε, ένα σημαντικό τμήμα των χρημάτων αυτών θα αφορούν την διαστημική ε, δραστηριότητα και θα πρέπει βεβαίως αυτή η επένδυση, αυτά τα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ε, η εμπλοκή των ενδιαφερομένων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως εξίσου σημαντική είναι η συνεκτικότητα που θα πρέπει να υπάρχει στα διάφορα προγράμματα. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαδικασία Αυτό μάλιστα αναφέρεται και διαφαίνεται σαφώς και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, σχετικά με, την, ε, με το περιεχόμενο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος. Είναι γεγονός ότι όπως είπε και η κυρία Νίμπλερ θα πρέπει να δοθούν όλα τα εχέγγυα στην, στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανία ότι θα μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Βεβαίως είναι είναι πλέον παγκοσμιοποιημένη η δράση και στον τομέα αυτό και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όχι μονάχα στα πλαίσια ε, των ε, συζητήσεων, των εμπορικών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι μόνο εκεί θα πρέπει να ληφθούν λοιπόν υπόψη τα στοιχεία αυτά, αλλά και στις γενικότερες ε, συμφωνίες και εμπορικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να δούμε επίση και τον σημαντικό τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς υπηρεσιών διαστήματος ε, ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη και ότι θα πρέπει να διευθετώνται και τα θέματα των προμηθειών, των διαγωνισμών και ενδεχομένως να λαμβάνεται και ρυθμιστική δράση όπου αυτή είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30. Ευχαριστώ. Και περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση, είναι η έκθεση Φράνκ Proust, Cars 2020 προς μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Το λόγο έχει ο εισηγητής Frank Proust για